Okay, colleagues. If could take... Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Να σας θυμίσω κάτι. Για σας που δεν ήσασταν εδώ χτες, θα γίνει ψηφοφορία. Στις 10 θα πάμε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και θα συζητήσουμε τη μετανάστευση θα συναντήσουμε τους νέους που συζητούν τη μετανάστευση και μετά θα συζητήσουμε την κοινή έκθεση με την ΑΦΕΤ για τη μετανάστευση. Ο κ. Διάς Δεμέρα είναι ο συγγητής μας. Η Ελένα Βαλένθιάνο και μετά από αυτό στις 11.30 θα γίνει ψηφοφορία στο, όσον αφορά το βραβείο Ζαχάροφ. Να σας υπενθυμίσω κάτι. Πρέπει να ειδοποιήσετε ποιος ψηφίζει από τις ομάδες σας για το βραβείο Ζαχάροφ. Και τα τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά μέλη. Αν έχετε αναπληρωματικά μέλη που θα ψηφίσουν την ομάδα σα, γνωστοποιήστε το στη γραμματεία πριν στι 11.30. Διότι μόνο αυτοί που θα είναι στον κατάλογο, στην ΑΦΕΤ, θα μπορούν να ψηφίσουν για το βραβείο Ζαχάροφ. 11.30 αυτό. Η αίθουσα είναι η 2Q2 για την κοινή αυτή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για χρηματοδότηση από τον υπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώση των ε, ΜΚΟ, συγγήτρια Έλλη Λάιν. Πίσω μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία παρακαλώ. Εκείνοι που κουβεντιάζουν εκεί πίσω μπορείτε να κάνετε ησυχία. Έλλη, Θε να πει κάτι για αυτό που θα ψηφίσουμε. Ναι, ευχαριστώ Λίντα. Ευχαριστώ όλους τους τις εισηγητές για το συνεργατικό πνεύμα που διέκρινε στις προσπάθειές μας, διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ τα μάλα λοιπόν. Εντάξει, ψηφίζουμε. Έχουμε πολλές συμβαστικέ, άρα εύκολα. Να ελέγξουμε καταρχάς ότι λειτουργούν τα μηχανήματα ψηφοφοριών, δοκιμαστική ψηφοφορία, πατήστε όποιο κουμπί θέλετε, δοκιμή κάνουμε. Πέρας. Δουλεύει όλα, μια χαρά. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 αποσύρεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας γίνει έλεγχος για την 33. η ψηφοφορία. Ο έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 40 αποσύρεται. Πάμε στη 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται, Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτονται, 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται, Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές. να ελέγξουμε την τροπολογία 50. Ξεκινά ηλεκτρονικός ελέγχος. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Α, Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτοτε. 54 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτοτε. 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. σημαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. σημαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 71 νομίζω ότι απορρίπτεται για την 71 τροπολογία 71 έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Ναι, πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια, Έλλη Σλάιν. Συνάδελφοι, σπάσαμε ρεκόρ. Η άλλη για την πρόσβαση στα φάρμακα έχει αναβληθεί, η άλλη ψηφοφορία. Οπότε θα, θα πάμε στο σημείο 12 στην αίθουσα 2Q2 για το υπόλοιπο πρωινό και το απόγευμα θα είμαστε πάλι εδώ. Στις 3 εδώ το απόγευμα. Αργότερα λοιπόν εδώ. Θα τα πούμε στις 10 στην 2Q2. Ευχαριστώ.